Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε την σύνοδο, την απογευματινή συνεδρίασή μας. Τα χθεσινά πρακτικά και τα εθετημένα κείμενα είναι διαθέσιμα. Ε, υπάρχουν κάποια σχόλια. Έχετε επιφυλάξεις όσον αφορά αυτά που ανέφερα. Δεν βλέπω να υπάρχουν, οπότε θεωρούνται τα πρακτικά εγκεκριμένα. Πάμε στην ημερήσια διάταξή μας. Συζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Επιτρέπουμε μία ώρα περίπου για αυτές τις συζητήσεις. Πρώτα σημείο, η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και συγκεκριμένα οι μαζικές εκτελέσεις και ο πρόσφατος θάνατος του blogger Σατάρ Μπεχέστη. Πρώτα απ' όλα, Ρωμίβα Ιρουέδα. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ιράν, στο Ιράν συνεχώς επιδεινώνεται. Πολλές περιπτώσεις βασανιστερίων, κακομεταχείρισης, αμελίες και θανάτους στο Ιράν έχουν καταγραφεί στον ο Μπεχέστη που ήταν 30 χρονών blogger συνελήφθη στις 30 Οκτωβρίου από την αστυνομία του διαδικτύου του Ιράν. Ε, έφτασε στο, φτάσαν στο σπίτι του και του κατάσχεσαν και διάφορα δικά του αντικείμενα και τους υπολογιστές του. Η οικογένειά του προσπάθησε να συλλέξει πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο Μπεχέστη και γιατί συνελήφθη από τι δυνάμει ασφαλεία και τι δικαστικέ αρχέ. Δεν του δόθηκε μέχρι 6 Νοεμβρίου απάντηση, όταν οι αστυνομικοί είπαν στην οικογένεια ότι ο μπλόγκερ πέθανε ε, ενώ ήταν υπο, τελούσε υποκράτηση. Οι αρχέ ε, δεν έδωσαν καμία εξήγηση για το θάνατό του. Γι' αυτό, σε αυτό το ψήφισμα, θέλουμε να ζητήσουμε άμεσως εξυχνίαση των συνθήκων για το θάνατο του Σατάρ Μπεχέστη ε, που ετελούσε υποκράτηση και να ζητήσουμε να διωχθούν οι υπεύθυνοι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και το δικαίωμα της οικογένειας που θέλει να εξηχνιάσει υπό ποιε συνθήκες πέθανε. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι η εκτέλεση στις 22 Οκτωβρίου 10 Ιρανών υπηκών ε, που θεωρήθηκαν χρήστες ναρκωτικών και θεωρούμε ότι δεν δικάστηκαν δίκαια και βασανίστηκαν ε, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Υπάρχουν πολλές περιστάσεις. Υποχρεωνόμαστε εκ νέου να ζητήσουμε από τις Ιρανικές αρχές να μην βασανίζουν πλέον τους φυλακισμένους, να μην τους κακομεταχειρίζονται και να μπορούν να έχουν πρόσβαση φυλακισμένοι στους δικηγόρους, της επιλογής τους και ιατρική περίθαλψη όταν αυτή απαιτείται. Ας μην ε, λησμονούμε ότι το Ιράν έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση των Πολιτικών ε, Δικαιωμάτων, Ιστικών Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, όλοι γνωρίζουμε ότι ε, το καθεστώς στο Ιράν δεν σέβεται τις υποχρεώσεις του έναντι του διεθνούς δικαίου και βλέπουμε ότι συνεχώς υπάρχουν προβλήματα ε, ότι ε, υπάρχουν βασανισμοί, διώξεις ε, και τα μέλη της, των μέσων ενημέρωσης τιμωρούνται και διώκονται. Ε, ένα, μια τέτοια απόδειξη είναι και ο θάνατος κατόπιν βασανιστήριων ε, του Ιρανού blogger Σατάρ Μπεχέστη ε, ενώ ελέγχθη ότι όλα θα πρέπει να επαληθευτούν παραμένει το γεγονός ότι υπάρχουν ε, ε, ντουζίνες πολεμίων του καθεστώτος οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξουν πλέον τέτοιες καταστολές. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα για το Ιράν. Μπορούμε να πούμε ναι ε, είναι μια χώρα με την οποία πρέπει να διαπραγματευτούμε ε, αντιλαμβανόμαστε πολλά πράγματα αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι την ε, βία και την σκληρότητα αυτής, ε, αυτού του καθεστώτος όπου αυξάνονται οι θανατικές καταδίκες και αντί ε, να μπορέσουμε να συναντήσουμε ε, τους ε, ε, δύο βαραβευθέντες με το βραβείο Ζαχάροφ δεν μπορέσαμε να φτάσουμε πουθενά. Πρέπει λοιπόν να γίνει μία έκκληση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δούμε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό και το Δεκέμβριο θα ήθελα να μπορέσουμε να εορτάσουμε το βραβείο Ζαχάροφ με τους δύο βραβευθέντες, τον κύριο Παναή και ε, ο οποίος κινδυνεύει να φυλακιστεί και τον συνβραβευθέντα του ο οποίος έχει κηρύξει απεργία πίνης. Ευχαριστώ. Και για ένα λεπτό ο κύριος Στίβενσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το φασιστικό καθεστώς του Ιράν έχει ε, χρησιμοποιήσει ένα ε, προπέτασμα καπνού και βλέπουμε ότι τις τελευταίες δέκα μέρες έχουν εκτελεστεί δέκα άτομα και αυτό προστίθεται στις 120.000 καταδικαστέντων που έχουν εκτελεστεί τα τελευταία χρόνια και έχω εδώ τον πρώτο μόνο τόμο από τα 20.000 ονόματα των αντιφρονούντων οι οποίοι έχουν εκτελεστεί. Είναι άλλωστε γεγονός ότι το κοινοβούλιο αυτό προσπάθησε ακόμη προενός μηνός να στείλει ε, προς ε, αυτό το κοινοβούλιο το, μια φιλική αποστολή ενώ ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ξαναστείλουμε φιλική αποστολή σε αυτό το φασιστικό καθεστώς ευχαριστώ τώρα για δύο λεπτά η κυρία, η κυρία Σάι Σαγιά ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η τωρινή κυβέρνηση στο Ιράν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της. Δεν πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε μόνο την ανησυχητική κατάσταση ε, για τον Σατάρ Μπεχέστη ο οποίος πέθανε στη φυλακή αφού είχε φυλακιστεί διότι ε, κατέκρινε στο facebook το ε, καθεστώς του Ιράν. Έχουμε διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για όλο και περισσότερες θανατικές καταδίκες και ε, πολλοί επισημαίνουν πόσο κακή είναι η κατάσταση στο Ιράν αλλά δεν βλέπουμε τη συνολική εικόνα δηλαδή ότι ε, ε, η, κυβέρνηση του Ιράν υποθάλπει την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και παραμένουμε αδρανείς παρακολουθώντας ε, ε, πώς αναπτύσσει το πρόγραμμα της πυρηνικών όπλων η κυβέρνηση του Ιράν ε, απειλώντας ότι θα εξαλείψει το κράτος του Ισραήλ και έστειλε και άλλα όπλα μέσω κρίσης ή στο Χαμάς. Γι' αυτό και ε, τα ίδια συμβαίνουν τώρα στο Ιράν που συνέβησαν και προηγουμένως στο Ιράκ σχετικά με την αντιπολίτευση εξού και είναι πολύ βασικό η Επίτροπος ε, Άστον να μπορέσει να ε, εφαρμόσει και να οξύνει τις ε, κυρώσεις, τις εμπορικές κυρώσεις κατά αυτού του καθεστώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό τώρα κύριος Μέρφη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο θάνατος του Σατά Μπεχέστη μετά από άγριους βασανισμούς, υποκράτηση και φυλακίστηκε μάλιστα για δράσεις κατά της ασφάλειας επειδή έβαλε κάποια πράγματα στο facebook. Αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Σύμφωνα με το Human Rights Watch, πάρα πολλοί άνθρωποι επειδή ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους βρίσκονται υποκράτηση κράτηση ή τραυματίζονται από βασανισμούς. Πάρα πολλοί ακτιβιστές επίσης έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και έχουν εκτελεστεί. Έξι άτομα το 2012. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Η καταστολή αυτή και η ακριότητα αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και σαν ε, άλλο σαν πρόσχημα για να γίνει στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Δεν ε, πρέπει να καταδικάζονται με κυρώσεις ούτε οι απλοί άνθρωποι στο Ιράν. Πρέπει να πετήσουμε το Ιράν να ελευθερώσει τους ε, πολιτικούς κρατούμενους και να καταργήσει τη θανατική ποινή. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά τώρα το λόγο έχει η κυρία Ούλαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, 22 Οκτωβρίου ο Σατά Μπεχέστη έγραψε στο blog του κάποια, ότι οι καταδίκες δεν γίνονται μετά από καμία δικαιοσύνη και με τρόπο που κανείς να μην μπορεί να αντιδράσει. Λίγο μετά ε, συνελήφθη, βασανίστηκε υποκράτηση. 3 Νοεμβρίου ε, πέθανε. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς. Διάφορες εκθέσεις λένε ότι πέθανε μετά από βασανισμούς. Αυτό δείχνει βάρβαρεο κράτος, το καθεστώς του Ιράν. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τις αρχές του Ιράνου να αρχίσουν και πάλι διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Σατά Μπεχέστη, όπως επίσης και σε όλους τους άλλους που έχουν υποφέρει από το σκληρό και βίο καθεστώς του Ιράν. Εμείς το έχουμε πει και ξαναπεί, δυστυχώς όμως δεν έχουμε πετύχει κανένα αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα αρχίζουμε με τους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Και πρώτος είναι ο κύριος Πόσελτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την πρωτοβουλία της ε, διεθνούς κοινότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους του Ιράν ο οποίος κάθεται πέντε χρόνια στη φυλακή για τον ίδιο λόγο για τον οποίο πέθανε και ο μπλόγκερ που μας απασχολεί και για τον ίδιο λόγο που διώκονται και ε, οι βραβευθέντες με το βραβείο Ζαχάροφ δικαιούνται να ε, εξασκήσουν ένα από τα βασικότερά τους θεμελιώδη δικαιώματα και το Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ένομο κράτος όταν δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα βεβαίως να διαπραγματευτούμε και να έχουμε ε, διότι το Ιράν είναι ένας από τους παλαιότερους πολιτισμούς της ανθρωπότητος αλλά θα πρέπει να φέρεται αντίστοιχα και ανθρώπινα έναντι προσωπικότητων οι οποίοι προσπαθούν απλώς να εκφράσουν ελεύθερα και ανοιχτά τη γνώμη τους. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ο Σαχτάρ είναι απλώ ένα παράδειγμα από την απώλεια ελευθερίας αντιπροσωπεύει την κοινωνία των πολιτών που εμπνέεται από την ελευθερία και τους επιτίθενται βάναυσα εδώ και καιρό. Ε, θα δούμε ότι υπάρχει έλλειψη κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πολεμήσει για τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Θα πρέπει να γίνει αμερόληπτη έρευνα, να διαπιστωθεί πώς πέθανε φυλακισμένος ο Σατάρ Μπεχέστη και να ενημερωθεί η οικογένειά του για τα αποτελέσματα. όπως επίσης και όσοι πήραν το βραβείο Ζαχάροφ ε, δεν τη χάνουν καλύτερη μεταχείριση και θα πρέπει να διορθωθεί κατά σοφά την κοινωνία των πολιτών. Ο κύριος Βοητσεκόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που επικρίνουμε το Ιράν για τις εκτελέσεις που πραγματοποιεί, αλλά αν δεν κάνουμε κάτι σοβαρό, κάποια σοβαρή δράση, το καθεστώς θα συνεχίσει αυτή την πορεία. Κάποια πράγματα δεν θα πρέπει να λησμονούνται. Το 1988, όταν ήταν υπουργό ο Μοσαβή, 30.000 πολιτικοί κρατούμενοι εξετελέστησαν εν ψυχρό σε λιγότερο από ένα τρίμηνο. Οι περισσότεροι ήταν οπαδοί του PMO. Ήταν ένα από τα χειρότερα εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας που δεν έχει ε, εκδικαστεί από κανένα διεθνές δικαστήριο ακόμα. Αν επενθυμίσω τη δύσκολη κατάσταση των Κούρδων τουλάχιστον έχουμε 23 πολιτικούς κρατούμενους που περιμένουν να εκτελεστούν. Ο Αλή Φασάρη Χουζάνγκ Ρεζάι, μεταξύ άλλων, Μπεχός Αλγάνι και γλόγμα Μαμοραντί. Ήρθε η ώρα να κινηθούμε. Πρέπει αμέσως να σταματήσει αυτό, να σταματήσουμε τις συναλλαγές με το Ιράν και να επιβάλλουμε πλήρεις κυρώσεις, ούτως ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα τους κοστίσει ακριβά. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Βερζά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε στο 7ο κατεπήγον για το Ιράν από την αρχή της θητείας μας. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τραγική σε αυτή τη χώρα και έχει το προνόμιο το θλιβερό η χώρα αυτή να βρίσκεται πρώτη όσον αφορά τις παραβιάσεις κατά κεφαλή. Από την αρχή της χρονιάς, έξι ε, καταδίκες με θανατική ποινή από τον Οκτώβριο, και το καθεστώς επιταχύνει τις εκτελέσεις ε, χιλίων καταδικασμένων ε, οργανώνοντας μια επιτροπή του θανάτου. Εμείς δώσαμε το βραβείο Σαχάροφ Ενσρίν Σοτουχτέ βρίσκεται σε απεργία πίνες. και ο Σατά Μπαχέστη έχασε τη ζωή του υποκράτηση. Έχουμε ένα ψήφισμα, ναι, αλλά οι εκτελέσεις αυξάνονται στη χώρα αυτή έχουν πολλαπλασιαστεί επί τέσσερα σε σχέση με πέρυσι. Δεν θα ήταν πιο χρήσιμο αντί για το ψήφισμα, αντί να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ δεν βρισκόμαστε μόνο για να έχουμε καλή θέληση. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Παλέσκης. Ευχαριστώ. Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόεδρε, στο Ιράν έχει επιδεινωθεί πρόσφατα τους τελευταίους μήνες κατά πολύ. Δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις φυλακίσεις και το θάνατο του Σατάρ Μπεχέστη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι το Ιράν δεν σέβεται τη Συμβασία Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Η πρόσφατη εκτέλεση πολλών Ιρανών πολιτών, οι οποίοι μάλιστα μπορεί να μην πέρασαν καν από δίκαια δίκη και η παραβίαση μεταξύ άλλων και του δικηγόρου για φαρπαναχή κτλ. Είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι ο καθεστώ αυτό δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει όμω εμεί να το απαιτήσουμε αυτό και να απαιτήσουμε διαφάνεια του δικαστικού και σοφρονιστικού συστήματο τη χώρα και μορατόριμο όσον αφορά τη θανετική ποινή ευθύ αμέσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα για ένα λεπτό, κύριο Στάνοκ. Πρόεδρε, με μεγάλη ανησυχία εδώ και χρόνια παρακολουθούμε την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να μην πω και την πολιτική κατάσταση στο Ιράν, που δυστυχώ επιδεινώνεται συνέχεια. Όπως δείχνει και το ψήφισμά μας, το καθεστώ του Ιράν είναι ένοχο για πάρα πολύ σοβαρέ παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάρα πολλοί άνθρωποι καταδικάζονται σε θάνατο χωρίς προηγουμένω να έχουν περάσει από δίκη Καταπιέζονται οι γυναίκε, οι μειονότητε, οι ράβοι, οι Κούρδοι κλπ. κλπ. Και δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Ο θάνατος του Μπεχέστη η υποκράτηση δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτη. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα διαθέτουμε για να βοηθήσουμε βέβαια το λαό του Ιράν κατά του καθεστώτος αυτού. Το, Ζαχάροφ, το βραβείο Ζαχάροφ, Τζαφάρο Παχάνη και Μασρίν Σοντουτέχ είναι βέβαια συμβολικό. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει νέα διπλωματική και πολιτική πίεση που θα πείσει το καθεστώς του Ιράν να μεταρρυθμίσει το δικαστικό και σοφρονιστικό του σύστημα για να βοηθηθούν οι πολίτες του οι οποίοι αξίζουν πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίε και κύριοι. Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία προσέλκυση προσοχή του Προέδρου. Κάτσε, έχω πολλού που θέλουν να πάρουν το λόγο. Σα παρακαλώ να είστε λίγο πιο σύντομοι και να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όλου. Πρώτα η κυρία Μπαλάρ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπω βλέπουμε το Ιράν κατάφερε να εκτελεί τους ανθρώπους με βιομηχανικό τρόπο, σε βιομηχανική κλίμακα. Η ιστορία του Σάχταρ Μπεχέστη είναι καθαρή απόδειξη αυτού. Να παραθέσω από το blog του. Χτες με απείλησαν. Απείλησαν να πούν στη μητέρα μου ότι σύντομα πρέπει να φορέσει μαύρα. Αν δεν κλείσεις το στόμα σου θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να το βουλώσεις και να μην δεις πληροφορίε αλλιώς θα στραγγαλίσουμε και θα παραμείνεις ανώνυμος. Κάθε μέρα ε, δεν σταματούσαν τα απειλητικά τηλεφωνήματα. Σαν Ιρανός λέω ότι δεν μπορώ να σιωπώ υπό το φως αυτών των δυστυχιών. Δυστυχώς σήμερα ε, θα έπρεπε να αποτίσουμε φόρο τιμής προς τους πολιτικούς κρατούμενους, προς τον πολιτικό αυτό και την οικογένειά του, αλλά χρειάζεται περισσότερα από να, να τους τιμήσουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος, ευχαριστώ Πρόεδρε, το ψήφισμα έχει σαν στόχο και τους πολίτες του Ιράν. Είναι ένα σαφές μήνυμα από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η φωνή του ελεύθερου κόσμου που ανησυχεί για τα τεκτενόμενα στο Ιράν και δημιουργείται και η ελπίδα ότι η ελευθερία, τα δικαιώματα των πολιτών θα ξαναέρθουν στους πολίτες του Ιράν. Θα ήθελα να πω στον Γάλλο συνάδελφο ότι επί σειρά ετών σε αυτή την αίθουσα και σε άλλες αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετούντο ψηφίσματα που αφορούσαν την ελευθερία και τα πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και τελικά έπεσε το τείχος. Δεν θα, θα πρέπει να έχουμε κάθε εμπιστοσύνη ότι είναι λογικό να αντιδρούμε, διότι έτσι βοηθούμε όλους εκείνους που υποφέρουν και είναι κάτι απαραίτητο. Η κυρία Γκούρμα έχει το λόγο, επόμενη. Αγαπητέ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, ε, λοιπόν, στι τελευταίε προεδρικέ εκλογέ του Ιράν η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν έχει επιδεινωθεί σταδιακά. Όλο και περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι ε, εκτελούνται. Άδικε δίκε, βασανιστήρια, περιορισμό θεμελιωδών ελευθεριών είναι μερικά παραδείγματα του πολλαπλασιασμού των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόσφατο θάνατο του Σαχτάρ Μπεχέστη είναι τραγική ε, υπενθύμηση τη καταστάσεω. Αυτό είναι κάτι που κρύβεται πίσω από τι εντάσει λόγω τη πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να δούμε με ποιο αποτελεσματικό τρόπο μπορούμε, με παραγωγικό τρόπο, να συζητήσουμε τι Ιρανικέ αρχέ. Βάσει τη διτή προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μπορεί οι κυρώσει να είναι αντιπαραγωγικέ και οι απλοί πολίτε να υποφέρουν παραπάνω. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρω τα νέα εργαλεία, όπω το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του γρήγορα. Να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ διαλόγου και κυρώσεων είναι κάτι απαραίτητο θέλουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Μιγκάλσκι έχει το λόγο. Πρόεδρε, θέλω να πω ότι ακούσαμε ότι από την ε, κυρία Βερζά ότι με τα ψηφίσματά μας δεν καταλήγουμε πουθενά. Ναι, αλλά είναι χρέο μας γιατί γίναμε ευρωβουλευτές και για να υιοθετούμε τέτοια ψηφίσματα γιατί και τα λόγια και οι λέξεις έχουν δύναμη απέναντι στο Ιράν. Ο κίνδυνος και η απειλή είναι διπλή. Πρώτον εσωτερική, στο εσωτερικό δηλαδή, όσον αφορά τους πολίτες του Ιράν, γιατί είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν σέβεται τους ίδιους του τους πολίτες. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με το Ιράν. Είναι μια χώρα που αποτελεί απειλή και για τους άλλους εκτός του Ιράν. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας λοιπόν. Εφόσον αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των Ιρανών, αγωνιζόμαστε και για τα δικαιώματα όλων να ζουν σε έναν ειρηνικό κόσμο. Ο κύριος Πρέντα τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο μπλόγκερ Σατά Μπεχέστη έχασε την ζωή του υποκράτηση. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επαναλάβει ξανά και ξανά και έχουμε καταγγείλει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Δημοσιογράφοι, bloggers, φοιτητέ, δικηγόροι, συνδικαλιστές ε, βλέπουν τα δικαιώματά τους να παραβιάζονται συνεχώς και τη ζωή τους να απειλείται. Θεωρούνται εχθροί του Ιράν. Ο Σέτα Μπεχέστη είχε το θάρρος να καταγγείλει τις καταχρήσεις του Ιρανικού καθεστώτος και τιμωρήθηκε με θάνατο τελικά υποκράτηση. Τον βασάνισαν, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι θάνατοι υποκράτηση στο Ιράν ε, δείχνουν ότι Τέτοιες ε, περιπτώσεις υπάρχουν πολλές. Θα πρέπει να τιμωρηθούν οι πέτοι. Εκ μέρους του ΕΛΚ εμείς στηρίζουμε τον ε, Γιαφάρ Πανάχη και την Ασρίμ Σοτούντεχ και ζητάμε την ελευθέρωσή τους. Για ένα λεπτό, η κυρία Καρέτου. Ευχαριστώ. Ο θάνατος του Σατά Μπεχέστη, του μπλόκερ αυτού, είναι κάτι σκανδαλώδες, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτα άλλο από το να εκφράσει τις απόψεις του ειρηνικά σε ένα μπλοκ. Το Ιρανικό καθεστώς λοιπόν παραβίασε πάρα πολλά πράγματα και έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Όπως ακούσαμε ήδη υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Τις καταδικάζουμε όλες. Πρόκειται για εγκλήματα. Ένα από αυτά τα εγκλήματα είναι και η μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στον μπλόκερ αυτό στην ε, φυλακή. Πρέπει να ερευνηθεί η περίπτωση και να τιμωρηθούν οι πέτοι. Πρέπει επίσης να υπάρξει ένα μορατόριο για να σταματήσουν οι θανατικές ποινές στο Ιράν που αυξάνονται συνεχώς τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να σταματήσουν και θανατικές ποινές σε βάρος ανηλίκων. Το Ιράν δεν σέβεται ούτε καν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών του. Ευχαριστούμε ο κύριος Γαλιτόρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όχι για πρώτη φορά και φοβούμαι ότι έχει για τελευταία. Συζητούμε για μια ακόμη φορά τη φρικτή κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν. Είναι μια χώρα οποία κυβερνάται όχι μόνο από δικτάτορες, αλλά πώς να το πω, από αγρίους. Δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο και δεν σέβονται το λαό τους, τον οποίο συλλαμβάνουν τον δολοφονούν εάν δεν συμφωνούν. Είναι μια χώρα που θέλει να λένε ναι οι πολίτες και άντρες και γυναίκες και αν δεν λένε ναι κινδυνεύουν σοβαρά. Η περίπτωση του Μπεχέστη είναι ακριβώς απόδειξη αυτού. Συνελήφθη, βασανίστηκε, δολοφονήθηκε. Και η είμαστε οικογένειά του, το, το μαζέψατε. Ήρθε η ώρα η διεθνή κοινότητα να γίνει σκληρή απέναντι στο Ιράν και να επιβάλλει κυρώσει που θα πλήξουν το καθεστώς να το υποχρεώσουν να σεβαστεί τουλάχιστον το διεθνές δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ πολύ. Το Ιράν έχει παραβιάσει ξανά και ξανά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο blogger ε, Σατά Μπεχέστη βασανίστηκε και έτσι έχασε τη ζωή του. Η ΦΑΤΑ, η αστυνομία του διαδικτύου δηλαδή του Ιράν, παρακολουθεί τον κόσμο, κάνει λογοκρισία. Τώρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο καθεστώς του Ιράν ότι δεν είναι δυνατόν να μεταχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο τους πολίτες του, να τους βασανίζει, να τους συλλαμβάνει, να τους καταδικάζει και να τους θανατώνει. Πρέπει να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη και πρέπει η συζήτηση αυτή να γίνει και να αποφασίσουμε για κυρώσει. Ευχαριστώ. την κυρία Πασέσκου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα της δημοκρατίας και γι' αυτό η υπόθεση του Ιρανού blogger με προβληματίζει όλος ιδιαίτερος. Η σύλληψη και ο θάνατος του ε, που έλαβαν χώρα υπό ύποπτες συνθήκες. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να πούμε γιατί εξέφραζε την άποψή του με δημοκρατικό τρόπο απέναντι στις αρχές. Τέτοιου είδου πρακτικές θα πρέπει να αποθαρρυνθούν παντιοτρόπως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να βρει τον τρόπο να ασκήσει πίεση επί των αρχών του Ιράν. Χρειαζόμαστε απελευθέρωση άμεση των πολιτικών κρατουμένων και διακριτική μεταχείριση κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων θα πρέπει να πάψει. Αναφέρομαι σε εκείνους που πήραν το βραβείο Ζαχάροφ που θα έπρεπε να μπορέσουν να παραλάβουν το βραβείο τους ε, από το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο αν το Ιράν θέλει να ξανακερδίσει εξοπιστία θα πρέπει να σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις όσον αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα. Τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Τσαρνιέσκι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, και εγώ έχω φρικιώ από αυτές τις εκτελέσεις στο Ιράν. Από 22 Οκτωβρίου με 14 Νοεμβρίου 100 άνθρωποι εξετελέστησαν πάνω από 120.000 εκτελέσεις από το 1979. Σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει αυτό το ρυθμό εκτελέσεων. Και έχουμε ε, μια αντιπροσωπεία φιλίας που θέλει να συσφίξει σχέσεις με το Ιράν. Είναι κάτι ε, ε, αμφισβητήσιμο. Και εκτελέστησαν πολλοί ως χρήστες ναρκωτικών. Οι περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι ανήκουν σε οργάνωση που επί τρει δεκαετίε προσπαθεί να φέρει τη δημοκρατία στο Ιράν. Πολλοί από τους, μερικοί από του φυλακισμένου του PMO είναι ο Ζανιάρ Μουράντι, Πλατήφη Μουστάφα Σαλίμι, αλλά και ο Χαμπίπ Σφάρη μεταξύ αυτών που εξετελέστησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ από τον Επίτροπο Ρεν να προβεί στα σχόλιά του, παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ για τα πολύ εύστοχα σχόλιά σας στην πολύ σοβαρή συζήτηση που είχαμε σήμερα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως ανησυχεί πάρα πολύ με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και η συνεχής καταστολή των πολιτικών αντιφρονούντων, των καλλιτεχνών, των blogger, των ε, ε, παικτών ε, και των μη κυβερνητικών οργανώσεων αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως καταδικάσει αυτή την κατάσταση ε, και αποδώσει το βραβείο Ζαχάρος σε δύο αντιφρονούντες ε, στην κυρία Σανταντέ και στον κύριο Αναχή. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα της προσιλώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η, ε, ο θάνατος του blogger Σαχάτερ Μπεχέστη είναι ένα παράδειγμα της ισχύουσας κατάστασης ε, και της καταστολής ε, των αντιφρονούντων στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως αντέδρασε, ζήτησε να υπάρξει μία πλήρης έρευνα στις συνθήκες ε, του θανάτου του και στη συνέχεια ανακοινώθη ότι γίνεται μία έρευνα και ότι οι υπεύθυνοι θα διωχτούν θα παρακολουθήσουμε από κοντά την κατάσταση διότι είδαμε ε, και ε, δίωξη ε, δικηγόρων που πρασπίζονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε προβεί σε διπλωματικά διαβήματα στο, στην Τεχεράνη επί του θέματος. Η εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινή μας ανησυχεί πάρα πολύ για το Ιράν γιατί έχουμε 338 εκτελέσεις ήδη εφέτος και αυτό ε, επιβεβαιώνει ότι το Ιράν είναι ένας από τους πιο συνήθεις χρήστες της θανατικής ποινής και πέραν, των δημοσί... πέραν αυτού οι δημόσιες εκτελέσεις είναι πολύ συνήθεις στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταχθεί σαφώς εναντίον της θανατικής ποινής και η κυρία Κάθριν Άστον έχει ε, εκδώσει την τελευταία της δήλωση στις 21 Οκτωβρίου καταδικάζοντας τις ε, ε, μαζικές εκτελέσεις των Ιρανών που καταδικάστηκαν για λαθρεμπορία. Ανησυχούμε συγχρόνως για την θέση των εθνοτήτων και μειονοτήτων στο Ιράν παρόλη την εγγύηση για ισότητα αντιμετωπίσεως Υπάρχουν πολλές μέθοδοι οι οποίες ε, ε, είναι αμφισβητούμενες και ζητούμε από το Ιράν να εφαρμόσει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και να καταργήσει τις διακρίσεις. Τώρα υπάρχουν, ε, υπάρχει η χώρα αυτή στον κατάλογο των χωρών που παραβιάζουν τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ε, την ε, ε, θέση του ειδικού εισηγητή Σαχέντ για το Ιράν και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε που μας μιλήσατε για αυτό το θέμα. Έχω έπτα ψηφίσματα